Okay, ladies and gentlemen, let's start. Ας ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Συγγνώμη που ακολουθήσαμε, που ξεκινήσαμε λίγο αργά, αλλά καλύπτεται το βέλιο από τρία ολόκληρα εκατοστά χιόνια. Φυσική καταστροφή. Και γι' αυτό καθυστερήσαμε. Κάποιες τροποποίησεις καταρχήν στη σειρά των ψηφοφοριών που είναι απαραίτητες λόγω των συμβαστικών λύσεων που επιτέθησαν από τους συντονιστές, ιδίως για τις προφορικές ε, τροπολογίες, η παράδοση της Επιτροπής μας είναι να επιτρέπουμε να γίνονται προφορικές τροποποιήσεις και πιστεύω ότι θα πρέπει να τη αυτή την παράδοση. Ξεκινάμε με την έκθεση «Γέτεν Μάκη» ε, ψηφίζουμε παραδοσιακά διανατάσεως χειρών και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες τώρα μετά για την πρωτοβουλία πολιτών που ίσως χρησιμοποιηθούν πιστοτικές κάλπες. Ξεκινάμε λοιπόν με την έκθεση. Γιατί μακή, τροπολογία 1. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 2. Υπέρ.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 Η 12 εκπίπτει. Εφόσον ενεκρίθη η 2, εκπίπτει η 2. Γι' αυτό πηγαίνουμε στην υπαριθμό 13. Okay. Amendment number 13. 13 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 14. Υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ. 17. Ψήφι για 17. Ψήφι Κατά. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Η 6 εκπίπτει 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. 18. Ψήφι υπέρ. Κατά. Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Και από εδώ και πέρα θα το κάνουμε ηλεκτρονικά. Γιατί έντος χρειάζονται αιώνες. So we're checking 18. για 18. Άρχεται. Ξεκίνησε η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρα στις ψηφοφορίες. 10-11 απορρίπτεται. Τροπολογία 8. 10-11 ήταν το αποτέλεσμα. Τροπολογία υπαριθμών 8 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίζεται. 19 ψήφι υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα. Μήπως μπορείτε να το ανακοινώνετε. 11-11, ναι, ναι. Δεν φαίνεται όμως ε, στο μαραφέτη μας εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τροπολογία 19, ψήφι υπέρ, ηλεκτρονικά. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά απορρίπτεται αποχές απορρίπτεται. 11 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση. Δεκατρία δέκα. Και πηγαίνουμε τώρα στην ψηφοφορία, στην έκθεση Γκουρμάη αλλά και Λαμασούρ για τις πρωτοβουλίες πολιτών. if adopted? If adopted, we Okay. So we start with amendment number Τροπολογία 104. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Απέριπτε. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην 113 τώρα. Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 της Επιτροπής Αναφόρων. Ψήφι Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 111 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 είναι ταυτόσιμη, δεν την ψηφίζουμε. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 10 της Επιτροπής Πολιτισμού καλύπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Πρώτο τμήμα καταρχήν. Α, συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την 115. 115, υπέρ. 115 υπέρ. 115 κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Επειδή συμφωνήσαμε ότι αυτοί που θα υπογράφουν θα πρέπει να καλύπτουν το 1 πέμπτο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 6 και αποφασίσαμε επίσης η Επιτροπή θα πρέπει να έχει 7 μέλη. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει και κάποια συνέπεια μεταξύ του αριθμού των χωρών και των ατόμων που είναι στην Οργανωτική Επιτροπή. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό, δεν είναι. Θέλετε να πάτε οι εισηγητές να κάνουμε κάποιο σχόλιο. <coughs> Όχι. Ψηφίζουμε, τι να κάνουμε. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Σοντάφ. Οι εισηγητές ε, δεν έχουν κάτι να πούν. <coughs> Τροπολογία 23. Ψηφίστηκε ήδη. 117. Ψήφι πάμε στην υπαριθμόν 11. Επιτροπής Πολιτισμού ψηφίτε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 119. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Δώδεκα είναι εγκρίνεται. Εκατόν εικοσιτέσσερα ψήφι υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 27 χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφιπέρ Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Το τρίτο τμήμα της 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 24. Ψήφι υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 13 ταυτίζεται. Προφορική τροπολογία του κ. κυρέλου Σαλόμ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. κάθε κράτος μέλος πρόκειται να αναλαμβάνει αυτές τις ενέργειες εκεί που λέει το, το, το, λέει για την ελάχιστη ηλικία. Η ελάχιστη ηλικία είναι αυτή που ορίζεται από το Κοινοβούλιο. Ε, το προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125, 125 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Ναι, της Λίμπη είναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτονται. 127 υπέρ. Κατά, αποχές, Απορρίπτονται. 25, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Το 14. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 129. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 Α, όχι, όχι, όχι. Η 27 της ε, Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών υπέρ, κατά, αποχές να απορρίπτεται. Η 26 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134. Υπέρ. Α, καταπίπτει. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Amendment number 28. Those members who are for, against. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Amendment number 30. Those... 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν σαράντα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίπε, Τριάντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πολιτισμού 17. Χωριστή ψηφορία. Οι συγκεκριτές έχουν αλλάξει γνώμη, δεν, θέλουν θέλουν χωριστή ψηφορία, αλλά την ψηφίζουμε όλοι μαζί. έγραφε χωριστή ψηφοφορία, αλλά ματαιώθηκε το αίτημα. Ναι. Πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα στις 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τριάντα Ναι, 31, υπέρ, Η 31 των συνεισηγητών. Υπέρ. Κατά. Το 31 ψηφίζουμε. Και πάλι ξαναψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πολιτισμού 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. Λίμπε. Πάμε στην 146 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Εδώ αυτό καταπίδει και πάμε στην 32. Θα έπρεπε να δούμε την 148 των πρασίνων, πρόεδρε. Α, συγγνώμη, ο πρόεδρος 148 ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Υπάρχει πρόβλημα γιατί έχουμε δύο μη εγγεγραμμένους αλλά μόνο ένας έχει ψηφίσει. Δύο-δύο από ε, συντηρητικούς ε, μεταρρυθμιστές. Α, εντάξει. Excuse me, excuse me for the mistake. Α, συμπαθάτε με για το λάθος, λέει ο πρόεδρος. Καλώς. Ok, από ό,τι φαίνεται, έχουμε έναν παραπάνω του ΕΛΚ. Μπας και μας προσμετρήσατε για σοσιαλιστές. Okay, ladies and gentlemen, let... Πρόεδρος, καλά κυρίες και κύριοι, επανερχόμεθα 148. Ξανά, καταμέτρηση των ψήφων υπέρ. Those members who are against. Κατά. Αποχές και απορρίπτεται. Και πάμε στο 32. Υπέρ. 32. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 20. Καταπίπτει. Λίμπε. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 λίμπε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τη Επιτροπή Συμφωνία 35 υπέρ κατά εγκρίνεται 151 είναι προφορική τροπολογία. Υπάρχει προφορική τροπολογία. 151 Ρούμπιχ προφορική αλλά απουσιάζει. Τι κάνουμε. Okay. Am I supposed to read it? Yeah, you should read it. Okay. Amendment 151 by Mr. Rubik, and I read it for you. Θα σας διαβάσω προφορική τροπολία μέσα σε 6 μήνες κατόπιν της θέσης ισχύ αυτού του κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να κοινοποιήσει ένα software λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά ε, σύμφωνα με τον ε, κανονισμό ε, και θα εξασφαλίσει επίσης την συντήρηση αυτού του software του λογισμικού. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Λίμπε. Συγχαρητήρια. Λίμπε. 37, 38, λέει ο πρόεδρο. Α, όχι. Αυτά. Ναι, θα το ψηφίσουμε. 37. Υπέρ, κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 38. Λίμπε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 152. Ε, Όχι, κατέπεσε και πάμε στο 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22. Calls 22. 153. Amendment number 153. There was 153. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 35. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Πολιτισμό 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αναφόρα 38, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πολιστικής, 23, υπέρ, κατά, αποχές, Α, απορρίπτεται. Λίμπε, 40, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 150, 4 υπέρ κατά υπέρ ξανά κατά αποχές απορρίπτεται 154 uh, all the others fall, uh, we have to vote on 37. Okay. So we go to... Και πάμε στο 37 των συνεζήγητων. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Yes, oral amendment or compromise amendment two. We go to go here. Okay. Compromise amendment number two. Συμβαστική υπαριθμών 2. Πάμε στην συμβαστική υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές 41. We go to petty 41 because all the other four. Αναφορών 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 43 ταυτόσιμη 167 those members 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Απολύτω. Σαράντα των συνεισηγητών υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Πολιτισμού. Okay, 41. των συνεισηγητών υπέρ, κατά, αποχές, γίνεται. Αναφόρον. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 συνεισηγητών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 της Λίμπε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπερθυμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. can be combined. Okay, 173. Those members who are for. 173 υπέρ. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτωση. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 48 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται 45 πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 182. Περ, κατά, απορρίπτεται. απορρίπτεται. Ε, αναφορών 47. Όχι, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, 182. Α, την ψηφίσαμε όμως. Άρα, πάμε στο 47 της αναφορών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 συνεισηγητών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν ογδόντα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αναφορών. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189. Υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 192. Απορρίπτεται. 46 συνεισηγητών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε. 50. Συνδυάζεται υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λίμπε 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λίμπε 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 Συνσηγητών. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 των συνεισηγητών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε. 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50, το πρώτο τμήμα έχει αποσυρθεί. Α, καταπίπτει. Καλό, με. Αναφορών 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 194. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λίμπε. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Συνεισηγητών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωται. Λίμπε, 56. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 συνεισηγητών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αναφόρων, 56. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 55, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. 199 είπα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 200 απόχες απορρίπτονται. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 της Επιτροπής Μουσείου Ελευθεριών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ εγκρίνεται. 59 καλύπτεται. 57. Τροπολογία 57 των εισηγητών. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 57. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59, Είναι ταυτίζεται με την προηγούμενη. Box 2, σημείο 5. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 60 λίμπε. Καλύπτεται. 203 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 57 κουτί 3 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Κουλτούρα 35. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 61. Η... Ταυτίζεται. Λίμπε 62. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59. Τροφορική τροποποίηση από τον εισηγητή κύριε Λαμασούρ. Εντάξει, δεν την ψηφίσουμε. Δεν τη διαβάσουμε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λίπε 3 Εκπίπτει. 60 των εισηγητών. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 204. Κατά. Ε, αποχές υιοθετείται. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Αφ καταπίπτει. Συγγνώμη. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 τους συνεισηγητές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 ε, 3 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 3 τους συνεισηγητές υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 66 καταπίπτει η πέτη 4 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Καλτ 1 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Καλτ 2 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68 4. Από τους συνεισηγητές. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Πέτη 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Από τους συνεισηγητές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Λίμπε 5. Όχι καταπίπτει αυτή. Προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών το εκτιμώντας 7 υπέρ. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Λίμπε 6. Α, όχι, καλύπτεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Α, υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Η 81 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 82. Υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 των συνεισηγητών υπέρ, κατά, άποχες, υιοθετείται. 8 από των συνεισηγητών υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 85 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 86 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται λίμπε 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Λίμπε 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 13, 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 των συνεισηγητών υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 11 των συνεισηγητών υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 12 των συνεισηγητών υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές υιοθετείται. 93 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Καλτ 8 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 του τους συνεισηγητές υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε Λίμπε 17 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Πάμε στη λίμπε 18. Πού ξαναρχίζουμε, κύριε Πρόεδρο. Λίμπε 19. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 15. Των συνεισηγητών. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείται. Λίμπε 20. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 16. Των συνεισηγητών. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Υιοθετείται. 91 υπέρ. Όχι, 99 διορθώνει ο πρόεδρος. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 απορρίπτεται. Αποσύρεται μάλλον. 5 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Τελική ψηφοφορία. Α, όχι, 103. 103. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Τι έγινε η προφορική ερώτηση στο άρθρο 2 σημείο 3. Η προφορική ερώτηση της, η προφορική τροποποίηση μάλλον της σοσιαλιστικής ομάδος. Την ψηφίσαμε και το αποτέλεσμα ήταν Εγκρίθηκε. Εντάξει. Τελική ψηφοφορία. Καταρχήν το έγγραφο της Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Ωραία, εγώ απέσυρα τη δική μου ψήφο. Πέρας ψηφοφορίας. 25-0. Τέλικη ψηφοφορία το, το νομοθετικό ψήφισμα. 25 υπέρ, η, καμία αποχή, καμία αντίθετη ψήφος, ομόφωνα. Και τελική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίστε όμως. Πέρα ψηφοφορίας. Πάλι ομόφωνα 25 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στους δύο συνεισηγητές. Και χρειαζόμαστε και να ψηφίσουμε για την εντολή που δίνουμε στους ε, δύο εισηγητές ηλεκτρονικά. Ας το κάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την εντολή των ε, εισηγητών, τελευταία, των εισηγητών, τελευταία ψήφος. Εντάξει. Πέρας. 24.00 εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mr. Mr. Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. President, Mr. President, I, Mr. President, I have a minor question. Έχω ένα ίσον θέμα, κύριε Πρόεδρε. Για την τροπολογία 191. Ενεκρίθη ή όχι. Απορρίφθηκε. Επειδή όμως ήταν μια ταυτόσιμη τροπολογία με την τροπολογία 190 και 190 εξέπεσε, δεν θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί 191. Εντάξει. Απλώς να βάλετε στα πρακτικά ότι δεν απερίφθη, απλώς ότι δεν ψηφίστηκε. Σύμφωνοι λέει ο πρόεδρος. Κύριε Χάφνερ. Μήπως μπορούμε να έχουμε λίγη ησυχία και να ακούσουμε τον κύριο Χάφνερ. Το άλλο μικρόφωνο δεν ε, λειτουργεί. Έχω ένα ερώτημα προς τον Πρόεδρο και στα έντιμα μέλη της Επιτροπής μας. Αν μπορώ να έχω την προσοχή σας για λίγο. επειδή έρχομαι από μια αλπική περιοχή της Ευρώπης και είχα πρόβλημα να έρθω. 8 ώρες ήμουν στο αεροπλάνο, δεν μπόρεσα να έρθω εδώ πέρα. Ο συντονιστής των Πρασίνων και συνεισηγητής για την Επιτροπή Αναφρών δεν υπήρχε κανένα πράσινο στην ε, Επιτροπή σας χθε. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να προσθέσω τώρα στο, στα πρακτικά την ε, συμβολή μας στη συζήτηση. Θα μπορούσα να το κάνω προφορικά, αλλά θα σας καταδαπανούσα τον χρόνο, αν υπάρχει δυνατότητα, να προσθέσω στα πρακτικά και την εξήγηση της θέσης των πρασίνων. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε την θέση των πρασίνων στα πρακτικά. Μπορείτε να την κάνετε γραπτά τη δήλωση αυτή. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ο Ινίγο. Δεν ήταν εδώ ο κύριος Χάφνερ χθε, αλλά το πνεύμα του διέπνεε όλη την Επιτροπή μας. Και σήμερα στις Βρυξέλλες μάθαμε ότι όλοι ζούμε σε μια αλπική κοινότητα. Τρία εκατοστά χιόνι και πλήρες χάος. Thank you, I just want to raise... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μέσερ και Σμιτ, θέλω να θέσω ένα ερώτημα μέσα στο ίδιο πνεύμα το οποίο μας ε, εμφορεί όλους μας. Φαίνεται ότι όλες οι ομάδες έχουν συμβάλει θετικά στην έκθεση αυτή, αλλά βλέπω στο τέλος του καταλόγου ψηφοφορίας ότι δύο ομάδες δεν συμμετέχουν στην προτινόμενη ομάδα διαπραγματευτών. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε μια πολιτική απόφαση ή σε κάποιο σφάλμα. <clears throat> Θα ήθελα όμως να θίξω αυτό το θέμα, διότι πιστεύω ότι οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές, όπως και η ομάδα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, που μπορούν να έχουν συμβάλει είτε θετικά είτε αρνητικά με τις τροπολογίες τους, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι μέσα στην ομάδα διαπραγματευτών μαζί με τους, τις άλλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος για την απουσία μας ή αν είναι κάποιο σφάλμα. Το έχετε ζητήσει επίσημα να είστε μέλο τη να είστε εκπρόσωποι στην ε, ομάδα διαπραγματεύσεως. Αυτό είναι η εξήγηση, λέει ο πρόεδρο. Πρέπει να υπάρξει μια επίσημη αίτηση και μετά θα συμπεριληφθείτε. Ωραία. Πρίμα. Uh, okay, what is the next on the agenda? The report by Mr. Duff. Okay, so shall we close this first part and... Έχουμε τελειώσει λοιπόν το πρώτο τμήμα, το τμήμα των ψηφοφοριών. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ταχύτητα με την οποία διεξήγατε, έχετε διεξαγάγει όλες τις ψηφοφορίες και το έκανε με χρόνο ρεκόρ ο Πρόεδρεύων. Ερχόμαστε τώρα στην επόμενη έκθεση, στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Ο Άντριου Νταφ μας παρουσιάζει μια νέα μορφή του σχεδίου του για την τροποποίηση του εκλογικού της εκλογικής πράξης του 1976. Ε, αυτό, αυτή η νέα πρόταση αφορά τρεις τροπολογίες οι οποίες είχαν κατατεθεί μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ε, μετά από μια συζήτηση στο συντονιστό ρεπτή. βάση αυτή τη συμβαστική λύση η οποία επετεύχθη στη συνέχεια, ο κύριος Νταφ κατέληξε σε ένα νέο σχέδιο του σχεδίου του. Θα δώσω καταρχήν λοιπόν το λόγο στον κύριο Νταφ και μετά στους βουλευτές οι οποίοι μπορεί να θέλουν να λάβουν το λόγο. Κύριε Ντουφ. Um, uh, Πρόεδρε. Μια στιγμή περιμένετε, λέει η Πρόεδρος. Άντριου. Μια στιγμή. Όλοι όσοι θέλουν να βγουν από την αίθουσα να βγουν τώρα, γιατί πρέπει να προσέξουμε τον συνάδελφο που θέλει να μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όλοι όσοι θέλουν να φύγουν, λοιπόν, να φύγουν σιωπηρά και όσοι επιθυμούν να παραμείνουν, ας παραμείνουν. Επίσης σιωπηρά. Ας ξεκινήσουμε. Α, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λέω ο κύριος Ντά. Θα ξέρετε ότι συζητήσαμε τα συστατικά αυτής της έκθεσης πολλές φορές. Κάναμε διαπαραταξιακές συζητήσεις και μου ζητήθηκε να μειώσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα στολίδια του. Δηλαδή τον κατάλογο των πραγμάτων που προτείνουμε να συμπεριλάβουμε στο πακέτο αυτό της εκλογικής μεταρρύθμισης. Μου ζήτησαν μάλιστα να μειώσω και το αίτημα περί συνέλευσης που προετοιμάζει την ε, διακυβερνητική που πρέπει οπωσδήποτε να συνταχθεί αν θέλετε, αν θέλουμε να περάσει αυτό το πακέτο της μεταρρύθμισης. Νομίζω ότι ακολούθησα τις επιθυμίες της Επιτροπής και υπέβαλα μία πιο ισχνή εκδοχή του κειμένου. Στην παράγραφο 2 θα δείτε ότι υπάρχει μια πρόταση για μια υπερεθνική λίστα για να εκλέξουμε 25 αναπληρωματικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. από μια πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια. Αυτή η πρόταση έχει επιβιώσει και είναι το απόσταγμα των προτάσεών μας. Αυτός ο κατάλογος θα αποτελείται από ένα τρίτο των του τουλάχιστον και θα είναι ισορροπημένο ε, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις ανδρών και γυναικών που περιέχει. Και προτείνω να είναι ημιανοιχτός προτιμησιακός κατάλογος, ούτω ώστε κανείς να μπορεί να, μπορεί να αποφασίσει για το κόμμα, όλη τη λίστα του κόμματος αν, που οργανώνει, οργανώνουν τα πολιτικά κόμματα ή αν επιθυμεί να πρημοδοτεί ένα συγκεκριμένο υποψήφιο. Στη δεύτερη περίπτωση, ένας μεμονωμένος υποψήφιος μπορεί λοιπόν να ανέβει σε αυτόν τον κατάλογο. Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της παραγράφου 3 είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε ένα μαθηματικό τύπο για την κατανομή των, 500, των 751 έδρων. Η αναδιανομή θα γίνει κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας και θα αντανακλά τις δημογραφικές αλλαγές και τα μεταναστευτικά μοντέλα που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη. Θα γίνει ένα συνέδριο, όπως γνωρίζετε, μαθηματικών στο Cambridge στο τέλος Ιανουαρίου που θα αποπειραθεί να δημιουργήσει μια συνένεση μεταξύ των μαθηματικών A γύρω από ένα μαθηματικό τύπο. Αν τα καταφέρουν, εγώ πιστεύω θα το καταφέρουν, τότε μπορούμε να συζητήσουμε εάν ο τύπος επί του οποίου θα έχουν συμφωνήσει είναι επαρκής για να εξασφαλίσει και μια πολιτική συνένεση. Το τρίτο στοιχείο στην παράγραφο 4 είναι η επανάληψη της πρότασής μας για το χρόνο των εκλογών, να μην γίνονται πια δηλαδή τον Ιούνιο, αλλά τον Μάιο, στην παράγραφο 6, ζητάμε από την Κομισιόν να αναθεωρήσει την οδηγία 93-109 που προσπαθεί να διευκολύνει την ψηφοφορία σε κράτη τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που διαμένουν ε, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγραφος 7 επαναλαμβάνει το μακρόπνο αίτημα του Κοινοβουλίου για το πρωτόκολλο του 65 για τα προνόμια και ασυλίες των βουλευτών που αναθεωρείται επίσης ως τμήμα αυτού του πακέτου. Στα παρατήματα επίσης θα δείτε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις της πράξης του 1976 που συνάδουμε τις προτάσεις του ψηφίσματος και στο δεύτερο παράδειγμα τις προτινόμενες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του πρωτοκόλου για τα προνόμια και τις ασυλίες των βουλευτών. Πιστεύω τώρα ότι με αυτή την έκθεση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στις τροπολογίες και στην ψηφοφορία, τόσο στην Επιτροπή, όσο και στην Ολομέλεια. Να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την νομιμότητα του Κοινοβουλίου λόγω της <coughs> νέας συνθήκης και όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και των θεσμικών οργάνων. στα πλαίσια της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει και η νέα συνθήκη. Περιμένω σχόλια από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Τρεις ε, συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Is there... yes, and shorts, yes. Is there anybody... Υπάρχει άλλος ο οποίος θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Φόξ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Άντζου Νταφ για την δουλειά που έκανε για αυτή την έκθεση. Σας παρακαλώ αυτοί που κάθονται πίσω μου να σοπάσουν, γιατί με ενοχλούν. Ευχαριστώ. Είναι βελτιωμένη αυτή η έκθεση σε σχέση με την έκθεση που μας είχε παρουσιάσει πριν από λίγους μήνες. Και οι πιο περίεργες ιδέες έχουν φύγει από το κείμενο. Χαίρομαι γι' αυτό. Η παράγραφος 2 της έκθεσης, δηλαδή η δημιουργία αυτού του υπερεθνικού καταλόγου, της υπερεθνικής λίστας, δεν μου αρέσει. Την απορρίπτω εντελώς αυτή την ιδέα. Η ιδέα επίσης ότι χρειαζόμαστε μία ε, Ευρωπαϊκή Εκλογική Αρχή που θα επιβλέπει τις εκλογές αυτές, θα εποπτεύει τις εκλογές, είναι περιττή. Και από πού προκύψω κάτω-κάτω αυτή η ιδέα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ζητήθηκε από κανέναν από κανένα φορέα να υπάρξουν επιπλέον 25 ε, βουλευτές. Η ιδέα ότι ο, οι λαοί που εκπροσωπούμε θεωρούν ότι αυτή είναι μια καλή ιδέα είναι παράλογο. Φαντάζομαι ότι πολιτικοί το σκέφτηκαν. Εδώ, η ελίτ των Βρυξελών, ε, αυτοί που ονειρεύονται το Μοσπονδιακό κράτος και δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τις ανησυχίες των λαών που εκπροσωπούμε. Θα καταψηφίσω λοιπόν αυτή την έκθεση όταν φτάσουμε στην ψηφοφορία και θα ήθελα, Άντριου, να διαγράψεις όλος διόλου την παράγραφο 2. Μα, αν το κάνεις, αυτό ε, η πρότασή σου ε, χτενίζει και βελτιώνει την πράξη του 1976. Μπορεί να έχουμε κάποιες διφωνίες, αλλά δεν είναι πρόβλημα όμως αυτές. Αν κρατήσεις την περιεθνική λίστα αυτή ε, και περάσει, ε, τότε θα, αποτελούσε μία, ένα ακόμα βηματάκι, ένα ακόμα λιθαράκι προς την Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Δεν θα μας άρεσε κάτι τέτοιο, φυσικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Νταφ που έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Μείωσε τις απαιτήσει στα πλαίσια του κειμένου. Είναι μια πιο μετριοπαθής εκδοχή από πολλές απόψεις ό,τι αφορά αυτόν τον υπερεθνικό κατάλογο. Το ΕΛΚΑ γενικά είναι υπέρ μια τέτοια ιδέα Για να απαντήσω στον κύριο Φόξ. Οι πρωτοβουλίες από κάποιοι προέρχονται. Δεν χρειάζεται να έρχονται από τη βάση κατά ανάγκη. Αν κάθε πολιτικό σύστημα ε, βασιζόταν στις πρωτοβουλίες από τη βάση, θα γινόταν τίποτα τελικά. Μπορεί κάποιες πρωτοβουλίες να προέρχονται από τις Βρυξέλλες, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν έρχονται είτε από τις Βρυξέλλες είτε από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Ο υπερεθνικός κατάλογος θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο για να συνδέσουμε τα κράτη της Ευρώπης όχι με ομοσπονδιακό ντε και καλά τρόπο, και να επιτρέψουμε ε, πολίτες από τη μία περιοχή της Ευρώπης να έρθουν σε επαφή με τους ε, άλλους πολίτες, ε, πολίτες που βρίσκονται αλλού. Ο μαθηματικός τύπος είναι ένας αλγόριθμος στην πραγματικότητα. Καλό θα ήταν να υπάρξει κάτι τέτοιο για να δούμε τι θα προκύψει από το συνέδριο των μαθηματικών στο Cambridge. Ευκταίο είναι να έχουμε μη πολιτικά αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή των εδρών. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ε, ενδυναμώνεται η αξιοπιστία του οργάνου μας. Δεν έχω πρόβλημα με τις εκλογές το Μάιο. Επίσης, ε, άτομα τα οποία ζουν μακριά από τον τόπο τους ε, να μπορούν να ψηφίζουν. Είναι επιθυμητό κάτι τέτοιο. Το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Αν σε κάποια φάση, σύντομα ας πούμε, συζητηθεί το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης ε, σε μια διακυβερνητική διάσκεψη, θα ήταν σημαντικό το θέμα της εκλογικής μεταρρύθμισης να συμπεριληφθεί επίσης ε, στην ατζέντα της διακυβερνητικής, γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται διαφάνεια και η λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ λοιπόν, λοιπόν τον κύριο Ντάφα. Ευχαριστώ. Και εγώ. Εν ονόματι των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ευχαριστώ τον Άντριου Νταφ για την προσπάθειά του για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και για το νέο του σχέδιο του κειμένου, το οποίο μας παρουσίασε και που μειώνει σε δύο βασικά, βασικούς τομείς της καινοτομίας, στο άρθρο 2 και το άρθρο 3, που φυσικά δημιουργούν πολλές πολεμικές και πρέπει να τα προσέξουμε όλους ιδιαίτερως. Για το άρθρο 3, το μαθηματικό αυτό τύπο. Συμφωνώ αυτό το σημείο να βρίσκεται στην πρόταση, στο κέντρο της πρότασης του Κοινοβουλίου, γιατί πρέπει το σύστημα μας να αλλάξει από αυτό το συνεχές ε, παρεδώσε και παζάρεμα στο Συμβούλιο για την αναδιανομή των εδρών. Φυσικά, το να εκχωρήσουμε στους μαθηματικούς τον, την εξέβρεση του μαθηματικού τύπου είναι μια προϋπόθεση ικανή αλλά όχι αναγκαία. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί μαθηματικοί τύποι και η επιλογή του καλύτερου τύπου είναι τελικά πολιτική και όχι των μαθηματικών και δεν τεχνική πρόταση. Η μειούμενη αναλογικότητα θα μπορούσε να εξασφαλιστεί με διάφορους τρόπους που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αναλογικότητα, μεγαλύτερη γραμμική μείωση κτλ. Τώρα, αν θέλουμε μεγάλη αναλογικότητα, δηλαδή ε, μεγάλη μετακίνηση εδρών από μικρομεσαίες ας πούμε χώρες σε μεγάλες, αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτήν την επιλογή στους μαθηματικούς. Οι μαθηματικοί μπορούν να μας βοηθήσουν να παρουσιάσουμε το πρόβλημα, να παρουσιάσουν ας πούμε δύο-τρεις επιλογές καθαρές. Από εκεί πέρα είναι θέμα πολιτικό το. Ποια λύση θα επιλέξουμε, ποια θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη. Γνωρίζουμε την παραβολη, τον παραβολικό τύπο, την ε, μέθοδο του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, δηλαδή αναλογικότητα συνέξη για όλους, ε, κάτι που μας εξασφαλίζει μεγαλύτερη αναλογικότητα. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να τονίσω. Επίσης, από πρακτικής απόψεως, επειδή χρειαζόμαστε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε πολιτικά με βάση αυτό που θα μας προτείνουν οι μαθηματικοί στο Cambridge, νομίζω ότι από διαδικαστικής απόψεως είναι λογικό να έχουμε προθεσμία για τις α, τροπολογίες επαρκή μετά το συνέδριο των μαθηματικών. Δηλαδή, θα γίνει το συνέδριο, εν συνεχεία μία συζήτηση εδώ και μετά τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τροπολογίες βάσει των αποτελεσμάτων ε, των εργασιών των μαθηματικών. Φυσικά, αυτό με κάνει να προτείνω να μας δοθεί επαρκής χρόνος, ούτως ώστε να συζητήσουμε τα αποτέλεσμα του συνεδρίου πριν ε, υποβάλουμε τις τοπολογίες. Δεύτερον, για το άλλο μεγάλο σημείο, το άρθρο 2, που αφορά την υπερεθνική λίστα. Με οδηγεί σε αντίστοιχο συμπέρασμα για τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτός ο κατάλογος του Νικοπέντε, ή μάλλον πέρα από την ουσία, έτσι, το θέμα είναι αμφιλεγόμενο, όπως ξέρετε από μεθοδολογικής απόψεως πρέπει να αλλάξει η συνθήκη. Όπως υπενθύμησε και ο Νταφ, έχουμε, απέναντί μας έχουμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ξεκινήσει μια μεταρρύθμιση α, της συνθήκης για το άρθρο 122 και την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι ένα σημείο κρίσιμο, αποφασιστικό για το μέλλον του είδους της διακυβέρνησης της Ένωσης. Εμείς στο Κοινοβούλιο κάναμε μια πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή μας και θα πρέπει να φτάσουμε σε μια θέση και να, γίνει, να ξεκινήσει μια συζήτηση με το Συμβούλιο. Όλες οι λύσεις μπορεί να είναι ανοιχτές. Μπορούμε να απορρίψουμε την αίτηση της απλουστευμένης διαδικασίας του 48-6. Μπορούμε να πούμε, πούμε ότι είναι πολύ μεγάλο το θέμα για να φτάσουμε στο 48-6. Μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Υπάρχουν διάφορες λύσεις. Πιστεύω ότι όλα αυτά μας κάνουν να περιμένουμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου πριν ε, κάνουμε μία πρόταση για μεταρρύθμιση της ε, συνθήκης ε, που συνδέεται με το θέμα το εκλογικό. Δεν έχει νόημα να ψηφίσουμε πριν αποφασίσουμε τι θέση θα έχουμε απέναντι στο Συμβούλιο για το θέμα της μεταρρύθμισης της συνθήκης. Για αυτούς τους λόγους ζητάω να καθορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα που μας επιτρέπει στην Επιτροπή να περιμένουμε το πέρας του συνεδρίου των μαθηματικών για το μαθηματικό τύπο, να καθορίσουμε μια θέση του Κοινοβουλίου για την πρόταση που υπάρχει επιτάπητος για τη μεταρρύθμιση της συνθήκης, ακόμη δεν ξέρουμε όμως ποια είναι αυτή ακριβώς, και που αφορά η πρόταση αυτή την οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ο πρώτος εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Άντριου Νταφ για την ε, ε, δουλειά του που ήταν συνεπής, ήταν αξιόλογη. Υποβάλαμε τις τροπολογίες μας και πρέπει να σας πω ότι παραμένει το θέμα μια πρόκληση. Γιατί θυμώ ότι μετά τι εκλογέ όταν συγκροτήθηκε σε σώμα αυτή η Επιτροπή, το είπαμε ότι θα πρέπει να βρούμε μια νέα προσέγγιση και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και να καταπονήσουμε την έκφραση της δυσπιστίας, δηλαδή την αποχή από τις ευρωεκλογές. Σε συνδυασμό όλα αυτά και με την εξεταζόμενη, μελετούμενη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος. Καλύτερα είπαμε τον Μάιο παρά τον Ιούνιο και σε άλλα με υπόψη και τα εθνικά χρονοδιαγράμματα. Άρα είναι σωστό το να γίνει ε, αυτή η πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο, ώστε να μην γίνονται Ιούνιο εκλογέ, αλλά να γίνονται νωρίτερα μέσα στον χρόνο. Σύμφωνα με το πρώτο σημείο των προτάσεων ΝΤΑΒ, όσον αφορά την νομιμότητα που θα προσδώσει το Ευρωκοινοβούλιο μια καινούργια ε, κατανομή των εδρών ανά χώρα. Επίσης συμφωνώ με τις προτάσεις του όσον αφορά τον συνδυασμό της ε, λίστας της Ευρωπαϊκής που θα πρέπει να συνδυαστεί με τις εθνικές λίστες. Το θέμα είναι ποιος θα αποφασίσει για τους 25. Είναι θέμα δημοκρατίας. Έχουμε που έχουμε αυτή την δυσπιστία του κόσμου, ξαφνικά να τους παρουσιάσουμε και ένα κατάλογο 25 προσώπων από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικά κόμματα. Ε, τι είναι αυτό θα πούνε. Άρα να δούμε πώς θα συνδεθούν αυτοί. με τον κόσμο. Προσοχή επομένω να μην χειροτρέψουν τα πράγματα με αυτή την ιδέα. Έχουμε πάντως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και έτσι είναι δυνατόν να υπάρξουν υποψηφιότητες για λίστες για αυτά τα κόμματα. Ε, και αυτά τα κόμματα είναι αναγνωρισμένα από τα θεσμικά όργανα. Και βέβαια τα κόμματα αυτά μπορούν και δικαιούνται να ορίσουν το ποιοι θα είναι οι αίρετοί τους εκπρόσωποι ε, για να μπουν σε μια τέτοια λίστα. Σας παρέπω στο το 191 και έτσι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση γενικότερα. Επίσης, συμφωνώ και με αυτό που είπε ο συνάδελφος Γκολτιέρη. Πρέπει να συνδυαστεί ακριβώ αυτή η μεταρρύθμιση του λογοσύστημα με την αναθεώρηση τη συνθήκη. Άρα στην θέση εφαρμογή της της πρέπει να εντάξουμε και αυτή την προβληματική και το Φεβρουάριο να παρουσιάσουμε, να προτείνουμε το όλο χρονοδιάγραμμα και να δούμε πώς θα επηρεάσει το πολιτικό γίγνεσθε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή την αναθεώρηση τη συνθήκη και μια γενικότερη μεταρρύθμιση αλλά και το εκλογικό σύστημα πρόεδρος. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Χέφνερ. Maybe Κάποιος θα μπορούσε... να φτιάξει αυτό το μικρόφωνο το οποίο δεν δουλεύει. Ίσως αν μιλήσω γερμανικά θα καταλάβει καλύτερα το μικρόφωνο και οι διερμηνείς. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Άντριου Νταφ, ο οποίος με μεγάλη επιμονή και συνέπεια έχει προωθήσει αυτό το θέμα και έχει επιμείνει στο θέμα αυτό. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να εδραιώσουμε βήμα με βήμα την υπερεθνική δημοκρατία και ήδη με το προηγούμενο σημείο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών έχουμε κάνει ένα πρώτο τέτοιο σημαντικό βήμα και έχουμε δημιουργήσει ένα πρώτο σύστημα μέσω του οποίου μπορούν οι πολίτες πραγματικά σε υπερεθνικό επίπεδο να εκφράσουν την άποψή τους και το εκλογικό δίκαιο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει τον υπερεθνικό χαρακτήρα των ευρωεκλογών και έτσι να υπάρχει η δυνατότητα να προωθηθεί η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα λοιπόν μιας λίστας η οποία είναι υπερεθνική, η οποία θα δώσει στους πολίτες δυνατότητα όχι μονάχα εθνικούς υποψηφίους να ψηφίζουν, αλλά και υποψηφίους οι οποίοι ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και θεωρούνται ότι είναι πραγματικά ε, έγκυροι εκπρόσωποι των ε, ιδανικών της Ευρώπης και των στόχων στην Ευρώπη, εμείς ως πράσινοι το θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ θετική πρόταση και γι' αυτό την υποστηρίζουμε. Την υποστηρίζουμε εδώ από πολύ καιρό και ιδιαίτερα τώρα την υποστηρίζουμε στα πλαίσια της έκθεσης του Andrew Duff. Έχουμε λοιπόν την ελπίδα ότι επιτέλους ίσως θα υλοποιηθεί κάποια, κάποια τέτοια λίστα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευφύες από την πλευρά του εισηγητή ότι ο κύριος Νταφ εστίασε την προσοχή του στο θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι μας δίνει πολλές, μας θέτει ενώπιον πολλών προκλήσεων το εκλογικό δίκαιο και ακόμα υπάρχουν πολλά για το εκλογικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν μας ικανοποιούν ιδιαίτερα. Υπάρχει παραδείγματο χάρη το θέμα με το, την, ε, ε, της επιλογής των υποψηφίων στα κράτη-μέλη. Πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι δημοκρατικός, όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται πάντα σε εκλογές. Έχουμε το γεγονός ότι υπάρχουν, ε, παραδείγματο χάρη, μέλη τα οποία έρχονται σε μία λίστα για τις ευρωεκλογέ όχι μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας αλλά μέσω μιας απόφασης κάποιων κομματικών οργάνων και μόνο. Αυτό δεν το θεωρούμε ότι είναι απόλυτα δημοκρατικό όταν δεν έχουν δυνατότητα οι πολίτες να ανθρωποποιήσουν τους εκλογικούς καταλόγους αλλά θα πρέπει να υποκύψουν, να αποδεχτούν έμεσα μυρολατρικά τις αποφάσεις πολιτικών εθνικών κομμάτων για τις ευρωεκλογέ. Η έκθεση του Άντριου Νταφ εστιάζει σε μερικά σημαντικά σημεία καταρχήν να γίνονται οι εκλογές το Μάιο και όχι τον Ιούνιο. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό και το υποστηρίζω ιδιαίτερα και σας υπενθυμίζω ότι ήδη είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό και στην, ε, ε, στα πλαίσια της έκθεσης του Άντριου Νταφ για τις ακροάσεις των Επιτρόπων. Είχαμε αποφασίσει ότι θα αποτελούσε μια μεγάλη βελτίωση στο χρονοδιάγραμμα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνεται νωρίτερα γιατί στη συνέχεια αυτό θα τη δυνατότητα να προχωρούμε στη διαδικασία κρόσης των επιτρόπων με πιο λυσιτελή τρόπο. Και εξάλλου το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, σε πολλά μέρη της Ευρώπης, στις σκανδιναβικές χώρες, ε, λείπει πολλοί κόσμοι σε διακοπές και αυτό περιορίζει και τη συμμετοχή στους, ε, στις ε, εκλογές. Εγώ τώρα για το θέμα του κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ε, συνέλευση, μια συντακτική συνέλευση ή αν θα πρέπει να αποδεχτούμε την ε, απλοποιημένη μέθοδο. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο θέμα αυτό τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Αλλά ο διάβολος υποκρύπτεται μεταξύ των λεπτομεριών πάντα. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση μέσα στην οποία να μπορούν και οι πολίτε να συμμετέχουν και η οποία θα δημιουργήσει πολιτική νομιμοποίηση. Αν τα συζητάμε ώρα και τα διαπραγματευόμαστε και κλεισμένο των θυρών και λέμε στου πολίτε να αυτό αποφασίσαμε, αυτό δεν μα δίνει περισσότερη νομιμοποίηση αλλά μειώνει την νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι μονάχα από πρακτικού λόγου λοιπόν αλλά και από συνταγματικέ θεωρήσει προκύπτει ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να γίνουν με συμμετοχή των πολιτών, επομένως να υποστηρίξουμε μια συντακτική συνέλευση, μια συνέλευση η οποία θα εξετάσει αυτό το θέμα, γιατί αυτό θα αυξήσει και την νομιμοποίησή μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. συναρπάζομαι από αυτά που μας προτείνει ο συνάδελφος Άντζου Ταφ πάντα γιατί έχει τόσο εύστοχη σκέψη και τόσο οξία αντίληψη και με μεγάλη ακρίβεια μπορεί να μας παρουσιάσει όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να σχολιάσω μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Γκουαλτιέρη το θέμα του μαθηματικού τύπου ή αλγορίθμου. Δεν είναι πάντα τόσο σε ένας τέτοιο τύπος. Δεν υπάρχει μία μαθηματική λύση για την ε, μειούμενη αναλογικότητα. Το θέμα είναι ποια είναι η αίτηση που θα θέσετε σε αυτό το συμπόσιο για την εξέβρεση ενός μαθηματικού τύπου. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς από τους μαθηματικούς να δώσουν μονάχα αντικειμενικές ε, λύσεις. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μαθηματικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να διατυπωθεί μαθηματικά το πρόβλημα το οποίο έχουμε να λύσουμε. Υπάρχουν πολλαπλέ λύσει οι οποίε μπορούν να υπάρξουν. Τι μπορούμε να ζητήσουμε, τι μπορούμε να πάρουμε από του μαθηματικού. Σω να μα δώσουν μια πλειάδα λύσεων οι οποίε θα είναι σαφέστερε ή αισθητικά πιο ικανοποιητικές, αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική επιλογή. Το κάθε κράτο ενδιαφέρεται περισσότερο για τον αριθμό των ε, υποψηφίων, των ε, εδρών στο Κοινοβούλιο και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Τρία θέματα θέλω να θίξω για την ε, σύγκληση μιας συνέλευσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έχουμε τον προπολογισμό και τη διαμάχη των προπολογισμών. Δεν μιλάω καν για την χρηματοοικονομική κρίση και εξάλλου έχουμε μόλις απορρίψει τον προπολογισμό του 2011. Δεν θέλω να ξεκινήσω μια συζήτηση για το αν το πράξαμε ορθώς ή λανθασμένα. Αλλά αν απορρίψουμε τον προπολογισμό και ζητήσουμε μια συνέλευση, τι εντύπωση θα δημιουργήσουμε γύρω από τα άτομά μας. Θα πούνε ότι έχουμε μια καθήλωση για την εξουσία και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Επομένως δεν συζητώ αν χρειάζεται η συνέλευση ή όχι, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ιδιαίτερα το περιραίον περιβάλλον για αυτή τη συνέλευση και να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Για τους μαθηματικούς τύπους κύριε Σαγράδας, εδώ θέλετε το εξή ερώτημα. Υπάρχουν μαθηματικοί οι οποίοι εργάστηκαν για το θέμα αυτό τους τελευταίους, τα τελευταία τρία χρόνια. Όλα ξεκίνησαν με το Συμβούλιο Υπουργών όταν θέλησε να υπάρξει μια φόρμουλα η οποία αντανακλά καλύτερα την ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε περισσότερο είναι η συνεκτικότητα. Βέβαια, άμα βάλει κανείς τα στοιχεία σε ένα υπολογιστή μπορούν να βγουν διάφορες λύσεις. Αλλά αν πούμε θέλουμε ευθύνουσα αναλογικότητα, μετά πρέπει να αποφασίσουμε τι μορφή ευθύνουσα αναλογικότητα θέλουμε για να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι συνεκτικό. Όχι στην περίπτωση της συνθήκης, όπως στην περίπτωση της συνθήκης του Άμστερνταμ, που λέει, λέμε εντάξει, βαρεθήκαμε, σας ακούμε, σας δίνουμε δύο άντρε παραπάνω και μετά έρχονται άλλοι όπως έτσι έχει και οι Ούγγροι που δεν είχαν σωστή εκπροσώπηση κτλ. Και η κάθε χώρα έρχεται και αρχίζει και διαμαρτύρεται. και λένε οι άλλοι ότι πρέπει να είναι εκτός ποσοστώσεως ο πρόοδο και έχουμε τώρα 751 βουλευτές και όχι 750. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε τώρα είναι πολύ καλά. Μπορώ να βασανίζω τους φοιτητέ μου να επινοήσω ερωτήσεις όπως πόσους βουλευτές έχουμε τώρα βάσει των διαφορών συνθήκων. Γιατί κάθε συνθήκη λέει κάτι διαφορετικό. Το πρακτικό βέβαια θέμα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ξέρω ότι ο Άντρου ήθελε το ταχύτερο δυνατό να προωθηθεί το θέμα αυτό, αλλά έχει δίκιο ο κ. Αν αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σοβαρά από μαθηματική έποψη, πρέπει να έχουμε ένα συμπόσιο και επί τη βάση αυτού να υποβάλουμε τις τροπολογίες μας. Γιατί υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία, ένα από τα οποία είναι αμφιλογόμενο για πολλούς η υπερεθνική λίστα και το άλλο είναι η φόρμουλα. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει σοβαρότητα και να έχουμε και μαθηματική σκέψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αναμείνουμε λιγάκι. Όλοι μας, όλους μας γοητεύουν τα μαθηματικά και οι φόρμουλες. Αλλά αν πούμε κάτι τέτοιο θα επανέλθει το το πρόβλημα του Συμβουλίου και της ε, ειδική πλειοψηφίας και θα μας κυνηγάει τις νύχτες ως βαμβούλας. Ευχαριστώ και δεν βλέπω να ζητεί άλλο το λόγο. Α, έχει το λόγο. Ναι. ναι, ναι πρόεδρε. Διαπιστώσαμε ότι έχουμε αυτή αυτή την, τη διάταξη που αφορά τους καταδίκους. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Από νομικής πλευράς θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κριτήρια, να δούμε τι ορίζεται ως παραδεκτό. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη, θα πρέπει να το δούμε καλύτερα. Να το δούμε καλύτερα και να διορθώσουμε αυτό το οποίο αναφέρεται στην πρώτη εκδοχή του κειμένου, γιατί και αυτό το θέμα έχει να κάνει με το τι προσδοκούν από εμά οι Ευρωπαίοι, οι Πρόεδρος. Ευχαριστώ και δώσω το λόγο στον Άντριο Ντάφ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το ιταλικό αίτημα και αναφορά όσον αφορά την διαγραφή εκείνων που έχουν εκτίσει κάποια ποινή έχουν τέλο πάντων καταδικαστεί σε ποινικό δικαστήριο θα πρέπει να το μελετήσουμε καλύτερα γιατί θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να τους δοθεί δυνατότητα να συμπληρώσουν τις προτάσεις μας και να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των αναφερόντων. Να σας πω τι πιστεύω ότι οι εθνικές πρακτικές σχετικά με τις ποινές αποστέρησης θεμελιωτών δικαιωμάτων ή των πολιτικών ελευθεριών ή πολιτικών δικαιωμάτων είναι, έχουν τόσο, τόσο μεγάλη ποικιλία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση. τα περισσότερα κρατημέλη αυτό που ισχύει είναι ότι άπαξ και έχει εκτιθεί η ποινή στη δική της ελευθερίας και αν έχει πληρωθεί η χρηματική ποινή, τότε αποκαθίσταται κανείς πλήρωση στα πολιτικά του δικαιώματα. Εγώ ως εισηγητής δεν προτείνω να κάνουμε αυτό το οποίο ζητούν με την αναφορά. αν στο χέρι μου θα τους εξηγούσα για ποιο λόγο δεν είναι τώρα να του καλύψουμε το αιτήμά τους. Πάντως, είναι ανοιχτή αναφορά και μπορεί οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής μπορεί να διατυπώσει μια αντίθετη άποψη. Τώρα όσον αφορά την κατανομή των εδρών, αυτή ε, ε, ο αριθμός 751 και αυτή η προσφυγή σε μαθηματικό θα πρέπει να εξαρτάται από αν υπάρχει συμφωνία και να δούμε τι εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν, τι επιλογές υπάρχουν και κατόπιν να το κρίνει αυτό η Επιτροπή μας. Όπως αναφέρθηκε από το συνάδελφο, υπάρχει βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλά στοιχεία πάνω σε αυτό, τα έχω μελετήσει όλα και... Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει οργανωθεί κάποιο είδου ιδεών brainstorming για να δούμε τι εναλλακτικέ υπάρχουν. Ας το δοκιμάσουμε. Ίσως το πείραμα αποδώσει, ίσως όχι. Και ίσως δεν βγει τίποτα από τη συνάντηση στο Κέμπριτζ. Και θα πρέπει να το ξαναζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Οπότε, το Συμβούλιο θα πρέπει να επανέλθει στην κλασική μέθοδο όπως μας είπε ο συνάδελφος Ράφα. Προσοχή όμως να μην ενεργήσουμε αντίθετα από τα όσα προβλέπει η συνθήκη για αυτή την φθήνουσα αναλογικότητα για τους 18 οι οποίοι θα πρέπει να εκλεγούν και να προσθεθούν στο σύνολο. Το πρόβλημα είναι δύσκολο, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να το λύσω. Βέβαια, να το συζητήσουμε. Να δούμε τι θα αποφασιστεί μετά αλλά στον Ρομπέρτο Καλτήρη έχω να πω ότι είναι σημαντικό το κοινοβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του και να αποφασίσει για το αν θέλει ή δεν θέλει την ε, μεταρρύθμιση και η αναβολή. Δεν είναι πιστική απάντηση και αντιμετώπιση του προβλήματος της αποχής. Και όλες τις επικρίσεις σε σχέση με την νοημοποίηση του Κοινοβουλίου. Είναι καθήκον μας να ανακτήσουμε αυτή την χαμένη εμπιστοσύνη και την αμφισβήτηση της νομιμότητας και να γίνει μια εκστρατεία για τις εκλογές που να αντικατοπτρίζει για όλο το πολιτικό φάσμα τη δουλειά μας. Βέβαια πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό στοιχείο και να μην έχουμε 27 διαφορετικές ε, εθνικές ή ακόμα χειρότερα υπάρχει ακού χαρακτήρα ε, πολιτικάντικη εκστρατεία αλλά να μπορέσουμε με αυτή την εκστρατεία να πείσουμε και να καλύψουμε και αυτούς που δεν καλύπτονται από τις εθνικές προεκλογές εκστρατείες. Και αυτό αφορά και τον Αμένα Βασίλειο. Και τους δικούς μου εκλογής που βέβαια δεν με ψήφισαν θέλουμε εδώ να τα συζητάμε. Βεβαίω πρόκειται για παλιά φεντεραλιστική ιδέα του να, του να μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια δημοκρατία που να ξεπερνάει τα κράτη-μέλη. Και η ιδέα φυσικά και έχει άμεσα να κάνει με αυτό το οποίο συζητούμε, τη μεταρρύθμιση του συστήματος. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι προσέγγισης βέβαια, για το, πόσο δημοφιλές και αγαπητό είναι το κοινοβούλιο. Πάντως, θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο εξατομικευμένη ούτως υπήν η εκστρατεία του ώστε να είμαστε πιο αναγνωρίσιμοι παντού πέρα από σύνορα και να ελκύσουμε και τον ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωση του τύπου. ως πολιτικές προσωπικότητες που να απολάβουν αυτή τη αναγνώριση και δημοφιλίας πέρα από σύνορα και πάνω από κράτη-μέλη. Επομένω το πρόγραμμα εκστρατεία όπω δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Καλά τα είπε ο κύριο Σόλτ. Έχουμε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία μπορούν να αναλάβουν την ε, δουλειά αυτή, δηλαδή να εντοπίσουν, να βρουν, να ορίσουν υποψήφιους για αυτή τη λίστα των 25. Μεγάλη ευθύνη βέβαια. Πολύ καλά τα είπα ότι έχουμε 10 τέτοια ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα επίσημως αναγνωρισμένα φαντάζομαι 5-6 ε, από αυτά λειτουργούν σε περιεθνική βάση. Επομένως, στα πλαίσια αυτής μας της προσπάθειας θα πρέπει και πάλι να μελετήσουμε το καθεστώς που διέπει τα κόμματα και φυσικά τα της χρηματοδοτησής τους. Διότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει και νομοθέτημα του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου που να κατοχυρώσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Προσοχή, όμως, για το τι θα κάνουμε με το άρθρο 48 παράγραφος 6 όσον αφορά τη διαδικασία της μεταρρύθμισης σε σχέση με τη μεταρρύθμιση την εκλογική. Υπάρχει εδώ θέμα πολιτικό, αν θέλουμε, να αναβαθμίσουμε την οικονομική διακυβέρνηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Διότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της νοημοποίησης. θεωρητικά δεν μπορούν να συνδυαστούν, να συγκυραστούν αυτές οι δύο μεταρρυθμίσεις ε, του στήματος με την αναθεώρηση της συνθήκης, διότι θεωρητικά είναι διαφορετικά ζητήματα. Και ο Τζερόλ και εγώ πάντως είμαστε υπέρ, αλλά όπως διαπιστώσατε, εγκαταλείψαμε την ιδέα και οι δύο, τότε θα πρέπει να γίνει κάποιο είδου ε, συνέλευση, ε, αναθεωρητική διάσκεψη, κάτι τέτοιο. Εκτός βέβαια και αν αποφασίσει σχετικά το Κοινοβούλιο εν ολομελία, οπότε θα ενημερωθεί φυσικά ο κύριος Φανρομπάη και τότε τότε για τη διακυβερνητική θα κρίνει ο κύριος Κάμερον και εσύ είναι αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και εμείς να έχουμε μια, ας την πούμε, συντακτική συνέλευση. Και τότε θα έρθει η ώρα να δούμε αν αυτό είναι εφικτό, αν αυτό είναι επιθυμητό, τι συνεπάγεται. Όλα αυτά τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Αρκετά είναι αυτά. Προς το παρόν, ε, ναι, σας αρκούν αυτά, εντάξει. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι συνοριστές θα συναντηθούν νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή την ε, μεθεπόμενη. Καλά, θα το συζητήσουμε τότε. Τότε θα το συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε. Όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε παράλληλα για όλα αυτά τα θέματα και όσον αφορά τη μαθηματική λύση και οι πολιτικές ομάδες προβληματίζονται, το συζητάνε εδώ και μια διετία, επομένως θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε για το ναι ή το όχι. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να γίνει η μεταρρύθμιση. Αν με καλέσουν οι σοσιαλιστές, ευχαρίστως να τους τα πω. και να, να, δούνε την, την αποκαλούμενη προοδευτική πλευρά του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς για αυτά που είπε ο Ρομπέρτο Γκαλτιέρη. Ο πρόεδρος ε, σας διένει με αυτό το γράμμα για να έχει τις απόψεις σας και δεχομένω τις ε, τροπολογίες σας. Η δεύτερη παρατήρηση, ξέρετε ότι στις 13 Δεκεμβρίου από τις 6 έως τις 7.30 το απόγευμα έχουμε μια εκτακτή συνεδρία και μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Πρώτη ανάγνωση θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου και αν έχουμε μια ε, σαφή εντολή μπορούμε να προχωρήσουμε. Και εφόσον θα γίνει αυτό το γεγονός το συμπόσιο στο Κέμπρις 27-29 Ιανουαρίου το ερώτημα Άντζου είναι πως πρέπει να επανέλθουμε μετά από το συμπόσιο, την 1η Φεβρουαρίου. Γιατί όλοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι. Μπορούμε να έχουμε πιο ήρεμα Χριστούγεννα και την 1η Φεβρουαρίου μπορούμε να συστήσουμε στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα έχουμε ήδη τα πορίσματα του συμποσίου. και μετά στη συνάντηση των συντονιστών νομίζω μπορείτε να καταλήξετε σε μια σόφρονα απάντηση. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό και έχουμε μια ακόμα έκθεση του Ανδρέα Νταφ ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού που αφορά τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2010 η Επιτροπή μας είχε εξετάσει το έγγραφο εργασία του Άντζου Νταφ όπου ανατέμει τη διαδικασία ακροάσεων των υποψηφίων επιτροπών που έγινε πέρσι και παρουσιάζει απόψεις για μια μεταρρύθμιση της διαδικασίας αυτής. Λόγω της θετικής υποδοχής της οποίας έτυχε αυτό το έγγραφο στη συζήτηση, ο εισηγητής μας, ο Άντζου Νταφ, έχει υποβάλει μια πρόταση τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου που παρουσιάζονται με την έκθεση αυτή για συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τον Άντριου Νταφ, αγαπητέ Άντριου Νταφ, να κάνετε μια εισαγωγή στη συζήτηση και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν ενδεχομένως να λάβουν το λόγο και να σχολιάσουν. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την ε, διόγκωση της ε, συμμετοχής μου στη σημερινή συνεδρίαση αλλά έχουμε επίσης συζητήσει και την προετοιμασία και την διαδικασία έγκρισης των ε, επιτρόπων προηγουμένως και εδώ βρισκόμαστε σε επίπεδο πρακτικών αποτελεσμάτων αυτών των συζητήσεων. Αυτό το οποίο επιζητούμε είναι να τροποποιήσουμε τους κανόνες διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κανονισμό και να ενσωματώσουμε τα συμπεράσματα τα οποία, στα οποία καταλήξαμε στις προηγούμενες μας συζητήσεις. Αν κοιτάξετε την έκθεση, στην τρίτη σελίδα του σημείου 9 της ημερησίας διάταξης, λέω στην πρώτη παράγραφο ότι η Επιτροπή μας μετά από την διαδικασία έγκρισης των Επιτρόπων είχε υποσχεθεί να τροποποιήσει τον ε, κώδικα διαδικασίας προτού υπάρξει τροποποίηση και της ε, δήλωση συμφερόντων των Επιτρόπων. Φυσικά όλα αυτά δεν αφορούν εμάς και μόνο, αφορούν και τον Πρόεδρο Μπαρόζο. αλλά μου είπαν ότι αυτή η εργασία είναι εν σειρμό. Συνεχίζεται και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και πάλι τη συζήτηση με την Κομισιόν. Σε σχέση με τις συγκεκριμένες τώρα τροπολογίες. Η πρώτη μου τροπολογία έχει σαν στόχο να καλύψει ένα χάσμα το οποίο υπήρχε μεταξύ της εκλογής του Προέδρου της Κομισιόν που γίνεται το Σεπτέμβριο και των ακροάσεων των ε, υποψηφίων επιτρόπων. Όπως είδαμε πέρσι, αυτό το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού χάσματος ήταν η απόφαση του Προέδρου να κατανείμει τα χαρτοφυλάκια στους υποψήφιους επιτρόπους αλλά δεν είχε την ευκαιρία να έλθει και να εξηγήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είχε αποφασίσει να μοιράσει έτσι τα χαρτοφυλάκια και στις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έθεσε τα αντίστοιχα ερωτήματα για το γιατί έγινε ούτως η κατανομή των χαρτοφυλακίων παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια αίτηση από μένα και την Επιτροπή μας ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση για το θέμα της κατανομής χαρτοφυλακίων από την πλευρά της Κομισιόν, δεν θέσαμε τέτοια ερωτήματα. Επομένως, η πρόταση που έχω στην πρώτη τροπολογία είναι ότι ο υποψήφιος πρόεδρος της Κομισιόν μάλλον ο εκλεγής πρόεδρος της Κομισιόν θα πρέπει να έλθει ενώπιον μια κοινή συζήτηση τη ε, συνέλευση των Πρόεδρων και τη ε, συνέλευση των ε, Πρόεδρων Επιτροπών για να εξηγήσει τι επιλογέ του. Αυτό είναι πιο λογική διαδικασία από αυτή που γίνεται όταν ζητάμε όλο το Συμβούλιο να έρχεται για τη συζήτηση ενθρονισμού της Επιτροπής. Ποτέ δεν έχει γίνει βέβαια αυτό, δεν έχουν έρθει ποτέ όλοι και ούτε θα μπορούσε κανείς να περιμένει να έρθουν όλοι. Πιστεύω όμως ότι είναι σημαντικό ο κ. Φαν Ρόμπεϊ να είναι παρόν στην Ολομέλεια όταν γίνεται αυτή η συζήτηση. Να είναι και οι τρεις πρόεδροι λοιπόν των βασικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόντες. Η τροπολογία 3 και κάποιε άλλες προσπαθούν επίσης να διευκρινίσουν το ρόλο των συντονιστών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αξιολόγησης των ακροάσεων. Νομίζω πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των συντονιστών, ιδίω εάν δεν υποχρεώνουμε το σύνολο των επιτροπών να συζητήσουν μετά από τις ακροάσεις σε σχέση με την αξιολόγηση που θα δώσει κάθε επιτροπή για κάθε υποψήφιο. Η τροπολογία 4 αφορά τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των επιτρόπων που είναι υποψήφιοι. Προς το παρόν αποστέλλονται την τελευταία στιγμή στις επιμέρους επιτροπές αυτές οι εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάνε για ένα πρώτο κοσκίνισμα σε μια επιτροπή η οποία μπορεί να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στις επιμέρους επιτροπές εάν δει κάποια ατασταλία ή τιμητική ατασταλία ή αν θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα σε σχέση με την δήλωση οικονομικών συμφερόντων των επιτρόπων, των υποψηφίων επιτρόπων. Αυτό νομίζω θα είχε περισσότερο συστηματικό χαρακτήρα και θα μείωνε την ε, ευκαιρία να υπάρξουν παραταξιακές μάχες σε σχέση με τον ακέραιο χαρακτήρα ή την ε, σωστή συμπεριφορά κάποιου επιτρόπου και θα ήταν και πιο ισοδίκαιο σε σχέση με τους υποψήφιους επιτρόπους. Στην τροπολογία 6 θέλω να δώσω περισσότερη διακριτική ευχέρεια σε σχέση με την επιλογή των γραπτών ερωτήσεων στις ε, επιτροπές. Πολλές φορές οι ίδιες οι επιτροπές είχαν εκφράσει την ε, δυσαρέσκειά τους γιατί δεν είχαν απόλυτη ελευθερία να επιλέξουν ερωτήσεις προς τους υποψηφίους που να αντανακλούν πλήρως τις πολιτικές προτεραιότητες. Και το τελευταίο ουσιαστικό σημείο είναι όλα αυτά αλληλένδετα βέβαια. Είναι η τροπολογία 10 όπου προσπαθώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της παρακολούθησης, της συνέχειας. Τι γίνεται αν μια επιτροπή ή μια συνδεόμενη επιτροπή σε μια ακρόαση δεν είναι ικανοποιημένη με τον υποψήφιο ή δεν είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας. Το 2004, όπως θυμάστε, υπήρξε μεγάλη σύγχυση για το τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Και αυτό επίσης δεν είναι ιδιαίτερα δίκαιο για τους υποψηφίους. Επιμένω λοιπόν να υπάρξει μία μοναδική μονάχα αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο, όχι μία από κάθε επιτροπή που συμμετέχει, ώστε να μην βρεθεί αντιμέτωπο με αλληλοσυγκρουόμενε αξιολογήσεις από την κύρια επιτροπή και τις συνδεόμενες επιτροπέ. Υποχρεώνουμε λοιπόν τις ε, επιτροπές οι οποίες συνδέονται σε μία ακρόαση και συμμετέχουν να καταλήξουν σε μία κοινή θέση. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρξει πρόσθετη διαδικασία για κανένα επίτροπο, υποψήφιο επίτροπο, χωρίς τη συμφωνία και του Προέδρου του Απερχόμενου Κοινοβουλίου και του Νέου Κοινοβουλίου. Το έγγραφο εργασίας είναι προσαρτημένο στην έκθεση, το έχουμε συζητήσει. Νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να το εξετάσουμε και πάλι, να το ξαναδείτε. Ευχαριστώ. Ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη ζήτησε το λόγο, αλλά είναι απόν, δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Ο επόμενο ομιλητή. Ο κ. Ταρσκόφσκι. Σύντομα, Άντριου. Κάποιε επιτροπέ και οι δικοί μα μεταξύ, μα, μεταξύ του, ε, δύο ή τρεις περιπτώσει, αποφάσισαν να επιλέξουν ένα εισηγητή. Δεν θα πρέπει να είναι κάνοντα αυτό για όλε τι επιτροπέ. Φυσικά είμαι προκατηλημένο γιατί εγώ ήμουν εισηγητή. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια σαφήνει εδώ. Τα πράγματα ήταν πιο απλά σε επιτροπές. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας. Ένας κανόνας. Ο ίδιος στις επιτροπές. Δηλαδή, ή να το έχουμε αυτό το πράγμα ή να μην το έχουμε. Ο συντονιστής των σοσιαλιστών, Ερίκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το θέμα αυτό έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Ο κύριος Νταφ έχει χρησιμοποιήσει όλη την εμπειρία που έχει. Όλα αυτά που συνέβησαν το 2009, όταν αξιολογήσαμε δηλαδή τους ε, επιτρόπους, αλλά και στο παρελθόν. Και παρουσίασε μία έκθεση για το πώς ε, λειτουργήσαν τον, το φθινόπωρο του 2009 αυτές οι ανακρίσεις, αυτές οι κοινοβουλευτικές εξετάσεις των υποψηφίων ε, ε επιτρόπων. Γενικώ πώς όλες οι προτάσεις του είναι πολύ λογικές και πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Νομίζω ότι έχει νόημα το να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Για να μην συμβεί ξανά και ξανά, να μην γίνει δηλαδή αυτό που συνέβη το 2009, δηλαδή να έχουμε να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ καθυστερημένα. Καλό είναι λοιπόν να μην συμβεί κάτι τέτοιο για να μην δυσκολευτεί και το πρόγραμμα του κάθε επιτρόπου και η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τις υποψηφιότητές τους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και η, αν πάμε τις εκλογές το Μάιο αντί και τον Ιούνιο, θα μας επιτρέψει όλη αυτή η διαδικασία να γίνει καλύτερα. Να λάβουμε υπόψη μας και τις διακοπές τις καλοκαιρινές και αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να ξαναρχίσουμε τις εργασίες στο Κοινοβούλιο. και όταν ε, συσταθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανωθεί το έργο των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με ομαλό τρόπο. Επίσης, η προσωπικότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι παρόν, παρούσα μάλλον στην, ε, στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει οι, οι αρμόδιες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές να εργαστούν τόσο ώστε να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις με αποτέλεσμα να, κάνουμε, να υπάρξουν κάποιοι συντονισμοί ούτως ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις στους υποψήφιους επιτρόπους. Δηλαδή, να ομαδοποιήσουμε τα θέματα αυτό έχει νόημα. Όπως επίσης οι επιτροπές οι οποίες δεν είναι άμεσα αρμόδιες και καθέλην υπεύθυνε να συμμετέχουν στην τελική αξιολόγηση, αλλά μέσα στα πλαίσια, πλαισιωμένες μάλιστα από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Εμείς λοιπόν θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε και κάποιες τροπολογίες ε, στην έκθεση DAF. Παρ' όλα αυτά, δεν, έχουμε κανένα βασικό, κανένα θεμελιώδες πρόβλημα με την έκθεση του κ. DAF έχει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ε, σε αδρές γραμμές μπορούμε να συμφωνήσουμε το περιεχόμενό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο ο κύριος Μέσερ και Σμιτ. Ευχαριστώ, συγχαίρω και τον κύριο Νταφ και το θαυμάσιο έργο του. Θυμάμαι σε μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών συζητήσαμε κατά πόσο ήταν σόφρον κάθε ακρόαση να καλύπτει το ίδιο χρόνο. Δεν ξέρω αν ε, συμφωνείτε για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί με σεβασμό για όλους τους επιτρόπους, εγώ δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να δίνεται ο ίδιος χρόνος για τη συζήτηση του Επιτρόπου Εξωτερικών Υποθέσεων με τον Επίτροπο Πολιτιστικών Θεμάτων. Είναι σαφές ότι έχουμε άνισα χαρτοφυλάκια, άνιση σημασίας και δεν θα ήταν και δίκαιο και για τους επιτρόπους αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλο χαρτοφυλάκιο να έχουν τον ίδιο χρόνο με τους άλλους. Ίσως θα μπορούσε λοιπόν να έχουμε δύο ακροάσεις για τις εξωτερικές υποθέσεις των Επίτροπων Εξωτερικών Υποθέσεων σε δύο μέρες. Μία συζήτηση υπάρχουν για εσωτερικά, για εξωτερικά θέματα. Υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μπορούμε λοιπόν με μεγάλη ευκολία να έχουμε δύο συζητήσεις των τριών ωρών για τους επιτρόπους με ευμεγέθη χαρτοφυλάκια. Δεν είναι δίκαιο λοιπόν για τους επιτρόπους να είναι όλα ταυτόσιμα και ομοιογενοποιημένα. Δεν είναι ότι τώρα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι θα έχουν πόσε ώρε στην ακρόασή του, αλλά τουλάχιστον να αφήσουμε κάποια ευελιξία για τι μελλοντικέ διαδικασίε. Ευχαριστώ. Κύριο Σεντάγκο. Συγχαρητήρια πάρα πολύ συναρπαστική και εμβριθή ανάλυση σα Με κάθε σεβασμό προς την ε, πείρα σας, τις γνώσεις σας. Είχαμε, έχουμε κάνει συναντήσεις ήδη. Και τι να σας πω για το κέμπιζο, αφού δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Χέφνερ. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι τόσο καλό ώστε να μην μπορεί να βελτιωθεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η οποία ε, προτείνει ο Άντριου Νταφ και ήταν πολύ χρήσιμο το ότι μας ε, έδωσε τις σκέψεις του για τις προηγούμενες ακροάσεις και τις προτάσεις του για βελτίωση αυτής της ε, διαδικασίας. Έχουμε νομίζω συζητήσει αυτά τα ζητήματα ήδη στην Επιτροπή μας στο παρελθόν και γι' αυτό δεν χρειάζεται να μπω σε βάθος και να συζητήσω λεπτομέρειες των ε, προτάσεων αυτών. Είναι σίγουρα σημαντικό να έχουμε περισσότερο χρόνο, να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για να έχουμε και περισσότερο χρόνο για να οργανώσουμε τις ακροάσεις των ε, επιτρόπων και κάτι το οποίο ξεφεύγει και από το πλαίσιο της ε, έκθεσης είναι το γεγονός ότι πολλά φυσικά εξαρτώνται από το να έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή το Κοινοβούλιο να απορρίπτει ένα συγκεκριμένο επίτροπο χωρίς να χρειάζεται να απορρίψει συμπούρμπουλο όλο το σώμα των επιτρόπων. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ καλύτερη δυνατότητα και είναι υποχρεωμένο το Κοινοβούλιο πολλές φορές να καταπιεί κάποιους επιτρόπους γιατί δεν θέλει να απορρίψει όλο το σώμα των ε, επιτρόπων. Αυτό λοιπόν θα ήταν μια πρόταση που θα ήθελα να έχει και περισσότερη υποστήριξη. Και πάλι ο Άντζελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα πρώτα τον Ραφαέλ. Ναι, ε, αυτό για τον ορισμό των εισηγητών είναι καλή ιδέα. και είχε αποδειχθεί αποδίδει και εγώ το είπα στην τροπολογία υπαρθυμών 5 στην πρώτη παράγραφο για εκεί και λέω ότι δύναται να γίνει ορισμός των εισηγητών και ορισμένοι πρόεδροι ορισμένων επιτροπών ζηλεύουν, ζηλεύουν και φθονούν την δόξα, τέλος πάντων, το κύρος και θεωρούν ότι πρέπει να καταπολεμήσουν οτιδήποτε τυχόν απειλεί ακριβώ τη θέση τους. Και επομένω, γι' αυτό νιώθουν ασφαλή και καταπολεμούν και τους εισηγητέ. Γι' αυτό και λέω λοιπόν, είναι δυνατόν να γίνει ορισμός και εγώ πάντοτε θα θα να γίνεται αυτό, να γίνεται ορισμός εισηγητών και όχι ε, κάποιοι πρώτοι να λαμβάνουν και τις ε, και τις εκθέσεις για τις τρεις ώρες. Τώρα συμφωνώ ότι ίσως είναι κάτι το πάρα πολύ βαρετό για ορισμένους υποψηφίου επιτρόπους και συνέβη αυτό. Και εγώ την ταλαιπωρία την τράβηξα, ήμουν σε κάποιες τέτοιες εκλογάσεις. Ε, βέβαια, άμα έχουμε τόσο πολλούς επιτρόπους, κύριος είδε πώς θα βγει αυτή η ώρα. δεν ωφελούν επομένω σε τρεις ώρες. Αλλά βέβαια ισχύει και το αντίθετο. Έχει διατυπωθεί άποψη ότι θα πρέπει να δίνεται το ίδιο χρόνο σε όλους τους ε, επιτρόπους και το πρεσβεύει αυτό και ο πρόεδρο τη Επιτροπής μου το έχει πει προσωπικά. Να μην διαλέγει το κοινοβούλιο, δεν διαλέγει εκείνο το ποιοι είναι σημαντικοί από του υποψήφιου επιτρόπου. και ο αρμόδιος για την εξωτερική δράση επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική θέση. Και σχετικά σας παραπέμπω στην τροπολογία 7. Να το συζητήσουμε. Ξανά. Τώρα όσον αφορά το timing για τις εκλογές, Έχουμε την πρόταση να μετακινηθούν εκλογές από τον ε, Ιούνιο πάνε το Μάιο και άρα και η Κομισιόν να ε, ορίζεται τον Ιούλιο και ο πρόεδρος Επιτροπής μπορεί κατά διάρκεια του καλοκαιριού να κάνει την ε, κατανομή των χαρτοφυλακίων Οπότε και οι ακροάσεις να γίνονται κατά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και όχι τον Ιανουάριο, όπως συνέβη την τελευταία φορά. Δεν γίνεται να τα αποφτάσουμε όλα πριν τις διακοπές και άλλωστε ο πρόεδρος, θα πρέπει να έχει το χρόνο να κάνει επαφές με τους 27 όσοι είναι τέλος πάντων. Όσους τους υποψήφιους επίτροπους που θα του προτείνουν ε, οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων. Πρέπει να έχει επομένω το χρονικό περιθώριο. Καταρχήν πάντως συμφωνώ ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Μέχρι σήμερα μάλλον. Φυσικά να μην καταλήξουμε να περάσει το δεκάμινο χωρίς να υπάρχει μια ε, επιτροπή η οποία να μπορεί να λειτουργήσει πλήρω. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για του ε, ευρωσκεπτικιστέ, αλλά κακό για του ε, φεντεραλιστέ. Τζέραλτ, ναι. όσον αφορά την ψηφοφορία ε, για τον κάθε επίτροπο χωριστά. Αυτό ορίζεται από την συνθήκη και δεν προτείνω να αρχίσουμε την διαδικασία της τροποποίησης αυτής της διάταξης. Ίσως το 2014 είναι ε, η πιο κατάλληλη στιγμή για να κινηθούμε προς μια τέτοια μεταβολή. Για προθεσμίες τώρα. Ίσως ε, ο κύριος Σέφερ ε, γνωρίζει, δεν, ξέρω. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Σεπτέμβριο το μεσημέρι δεν ακούστηκε η ημερομηνία. Είχε και το το μικρόφωνο. Ε, Άντριο, ευχαριστούμε. Έχουμε τον κύριο Μίτεκ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει η Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει να γνωμοδοτήσει για αυτές τις προτινόμενες τροπολογίες τον εσωτερικό κανονισμό. Με βάση το σημείο 21 της νέας συμφωνίας πλαίσιο προβλέπεται αυτή η δυνατότητα όταν ο εσωτερικός κανονισμός θα επηρεάσει τις διαθεσμικές σχέσεις, κάθε φορά που τις επηρεάζει. Και ακόμα και όταν μιλάμε για τους υποψήφιους επιτρόπους και, τους, και τον υποψήφιο πρόεδρο της Επιτροπής, μιλάμε για τις διαθεσμικές σχέσεις. Δεν θα σχολιάσω τις προτινόμενες τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να εκφράσω την ευνομοσύνη της Κομισιόν για τη δουλειά του Κοινοβουλίου, δηλαδή ένα προβληματισμό εκ των υστέρων για τη διαδικασία των ακροάσεων. Εκτιμούμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Νταφ, το ενδιαφέρον κείμενο του Απριλίου που συνέταξε και την έκθεση, και την έκθεση που μας παρουσίασε σήμερα και που εξετάζουμε σήμερα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο τελευταίος ε, λόγος τον κύριο Ντάφ. Σωστό είναι αυτό που λέει η Επιτροπή, ότι πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις στην Επιτροπή για το θέμα αυτό και να συμπεριλάβουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Μας υπενθυμίζει πολύ σωστά την ε, Συμφωνία Πλαίσιο επίσης αλλά άτυπα συζήτησα όλα αυτά τα θέματα και με τον πρόεδρο Μπαρόζο και με τον αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς. Άρα γνωρίζουν τις προτάσεις που κάνω. Απλώς πρέπει να προβλέψουμε μια συζήτηση με τον, ε, υποψη... με τον Αντιπρόεδρο και Επίτροπο κ. Σεύκοβιτς κατά τη συνέχεια της όλης διαδικασίας εξέτασης του πακέτου. Πρόεδρος. Χθες είδαμε ότι έδειξε ανοιχτό πνεύμα και διάθεση για να συζητήσει μαζί μας και μας είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να επανέλθει και να συζητήσει μαζί μας. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάναμε. Να επαναλάβω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Η προτινόμενη ημερομηνία είναι η 16η Δεκεμβρίου μεσημέρι. Και στις 30 Δεκεμβρίου θα έχουμε, στις 13 Δεκεμβρίου μάλλον, θα έχουμε από τις 4 μέχρι τις 5.30 μία έκτακτη συνεδρία στο Συντονιστό, 6 με 7.30 μάλλον, την 31 Ιανουαρίου, 1η ε, και 2 Φεβρουαρίου έχουμε την ε, τακτική συνεδρίαση της ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ που υποστήριξατε την πρωτοβουλία των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο, την κυρία Γουάλης, τον κύριο Χέφνερ για την βοήθειά τους. Γιατί χάρη σε αυτή την συνεργασία οι συντονιστές έκαναν καλή δουλειά. Θα, θα σας ξαναδώ λοιπόν ε, στις 13 Δεκεμβρίου.